good that we have to be punctual. I hope to be. So, ladies and gentlemen, we are now uh, switching to a point. Και τώρα περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Ισότητα των φίλων στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται για κοινό σημείο με την Επιτροπή ΦΕΜ βάσει του κανόνα 55. Ε, Αντιπρόεδρος... Θα συμπροεδρεύσω λοιπόν με την κυρία Μπάρβαρα Ματέρα, αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΦΕΜ. Έχουν κατατεθεί 339 τροπολογίες ε, για αυτή την, το σχέδιο έκθεσης. Και τώρα εδώ θα συζητήσουμε ε, όλες αυτές τις τροπολογίες. Έχουμε όμως μία ώρα στη διάθεσή μας μόνο. Πρώτα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Φορέντζα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εξ μου και εξ ονόματος της κυρίας Μπιόρκ που είναι εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Γυναικών και που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα να ευχαριστήσω καταρχήν τους συναδάλφους, γυναίκες και άντρες, ε, τους κοιόδης εισηγητές για αυτή την κοινή έκθεση Ίντα Φαμ. Ευχαριστώ την Μπάρμπαρα Ματέρα, την κυρία Νό, ε, Νόκλ, την κυρία Γιούτο, την κυρία Τρουσέσκη από την Επιτροπή ΦΑΜ και την κυρία Σάιφη, Ροντρίγκε Πινιέιρο, Κάριμ Άουτο από την Επιτροπή Ίντα. Και τέλος ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο στο προσχέδιο έκθεσης για τη δουλειά που έκαναν, για τις οπολογίες που παρουσίασαν που όπως ακούστηκε πριν από λίγο είναι 336 ούτε λίγο ούτε πολύ. Κάθε πολιτική ομάδα του Κοινοβουλίου παρουσίασε ένα τμήμα των τροπολογιών που λάβαμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το θέμα της προοπτικής της ισότητας των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες. Ξέρουμε ότι για τα θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο, το Κοινοβούλιο είναι συχνά διαιρεμένο. Από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν, ένα μεγάλο τμήμα αυτών, ε, νομίζω ότι βελτιώνουν το πρώτο σχέδιο έκθεσης που παρουσίασα εγώ μαζί με την κυρία Μπιόρκ. Πολλές από τις τροπολογίες δείχνουν μια ευαισθησία στο θέμα της ισότητας των φύλων, πρέπει να το πω αυτό, ακόμα και όταν αυτή η ευαισθησία εκφράζεται με μια τελείως διαφορετική πολιτική άποψη, πολιτικό προσανατολισμό από τη δική μου. Αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια διαπαραταξιακή ευαισθησία για το θέμα της ισότητας των φύλων και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή δουλειά για να φτιάξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Ένα τμήμα των τροπολογιών που κατατέθηκαν προσανατολίζονται στο να εντάξουν την πρόπτικη της όδες των φίλων στις εμπορικές συμφωνίες. Εμείς θέλουμε να υπάρχει δεσμευτική ένταξη της διάστασης του φύλου ε, και της ότας του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες, ε, όπως επίσης και στην αξιοπεπή εργασία, στην πρόσβαση στην υγεία σε όλους, για όλους. Και εδώ συμπεριλαμβάνω και την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για το θέμα της πρόσβασης στην τροφή, στο νερό και σε ένα καθαρό περιβάλλον οτιδήποτε επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, και εδώ υπενθυμίζω ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών είναι ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ε, μη δασμολογική ποσόστοση. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εκεί εδράζεται η ευημερία των ανθρώπων εδώ στο, σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι μια δουλειά που τη συνδέω με μια άλλη έκθεση που έκανε η άλλη συγγήτρια και που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου του 2016 στην ε, Ολομέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες. Θα πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια στο κείμενο, όχι μόνο να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα, 100% ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να ενισχύσουμε την διάσταση του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες. Προσπαθώντας να καταστήσουμε δεσμευτική αυτή η διάσταση στις εμπορικές πολιτικές της Ένωσης. Μιλάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα γυναίκα των γυναικών. Να είναι δεσμευτικά. Εγώ και η κυρία Μπιόρκ πολλές φορές τονίσαμε ότι οι πολιτικές διεθνούς εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου. Υπάρχει και μια έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στην ε, Επιτροπή Ίντα, την οποία την έχουμε συζητήσει πριν από λίγο καιρό και το λέει ακριβώς αυτό. Εμείς όμως δεν ξεκινήσαμε μόνο από αυτό το οπτικό, την οπτική γωνιά. Ε, ήρθαμε και σε επαφή με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και μετά από αυτή την επαφή ε, ενισχύθηκαν οι πεπιθήσεις μας και οι απόψεις μας. Δυστυχώς, πολύ συχνά συνάδελφοι και σκιώδεις ε, εισηγητές δεν ε, ήρθαν στις συναντήσεις και χάσαμε μια ευκαιρία να εμπλουτίσουμε με τις απόψεις τους την έκθεση. Υπάρχουν διάφορες εμπορικές ε, πολιτικές ε, και θα έρθουν και πολλές άλλες ακόμα. Ε, εκεί πρέπει σε όλες αυτές να λαμβάνουμε υπόψη μας τη διάσταση του φύλου. Στην Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής για πρώτη φορά υπάρχει ένα κεφάλαιο για το θέμα της ισότητας του φύλου. Εδώ ευχαριστώ την εισηγήτρια που είναι εδώ, που είναι η κυρία Ροντρίκη Σπινέιρο. Αυτό είναι μια κατάκτηση πολύτιμη και νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για περισσότερες ε, κατακτήσεις για να μπουν ε, τα θέματα του φύλου στις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία του θέματος αυτού. Παράλληλα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα θέματα του φύλου δεν είναι ένα θέμα, αλλά μια προσέγγιση. Μια προσέγγιση που θα πρέπει να αφορά όλες και όλα τα σημεία της ε, πολιτικής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι πρόκληση, αλλά είναι στόχος. Υπ' αυτή την οπτική γωνία θα θέλω να εργαστώ επί της έκθεσης αυτής μαζί με την κυρία Μπιόρ. Την ε, Παρασκευή θα γίνει μια πρώτη συνεδρίαση σκιωδών εισηγητών και ευχαριστώ ακόμα μια φορά όλους για την προσπάθειά τους και ευχαριστώ ακόμα όλους όσους συμμετείχαν στην ε, εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ε, Ευχαριστώ. Τη, συνάδελφη, τη συνάδελφο. Και εγώ να σε ευχαριστήσω για την δουλειά σας, για την ανταλλαγή email, για τις συναντήσεις και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές με τους κοιόδης εισηγητές στο μέλλον για να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό. Θα ξαναπάρω το λόγο ως κοιόδης εισηγήτρια του ΕΛΚΑ. Δεν θα δώσω τώρα το λόγο στον εαυτό μου, όμως, αλλά στη συνάδελφο Σαΐφη. Συγγνώμη, η κυρία Σαΐθη. Δεν, να είναι, θα μπορούσε να είναι, παρούσα, να είναι εδώ, οπόμενος ο κύριος Σαντιάγκο Φίσας θα την αντικαταστήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μιλάω στο όνομα της ε, συναδέλφου κυρία Σαΐφη. Ευχαριστώ πολύ τις συγγήτρες για τις σημερινές παρουσιάσεις. Ο ΕΛΚ έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες για αυτό το σχέδιο έκθεσης προκειμένου να υπενθυμίσουμε τις θέσεις μας πάνω σε διάφορα θέματα. Συμμεριζόμαστε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκφράζεται στην έκθεση για την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου και της ισότητας ε, θα ε, ε, έχει ως αποτέλεσμα να επιφορηθούν όλοι από την εμπορική πολιτική. Έχουμε επίσης προσθέσει μία αναφορά, όπως και άλλοι συνάδελφοι, στην μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ε, συμμετοχή των γυναικών και τις σχέσεις τους με τις εξαγωγές. Ζητάμε η ισότητα ανδρών γυναικών να, υπό... να λαμβάνεται υπόψη στις εκτιμήσεις επιπτώσεων το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της ισότητα ανδρών και γυναικών, όπω και άλλα ε, εμπορικά ε, εργαλεία που ε, ζητούν, απαιτούν την υπογραφή και επικύρωση διαφόρων συμβάσεων που αφορούν την ισότητα ανδρών και γυναικών. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο ΕΛΚ δεν είναι υπέρ των δεσμευτικών διατάξεων σε ό,τι αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών στις εμπορικές συμφωνίες. Η ισότητα των φύλων πρέπει να προσεγγιστεί διαφορετικά. Ο ΕΛΚ δεν ε, συμφωνεί με την συμπερίληψη κεφαλαίων συγκεκριμένα για τη διάσταση του φύλου σε εμπειρικές συμφωνίες. Θα μπορούσαμε σε πρώτη φάση να εξετάσουμε την αναθεώρηση της συμφωνίας με τη Χιλή και ενδεχομένω να προσθέσουμε κεφάλαιο. Τότε θα είναι μια πρώτη προσπάθεια, μια δοκιμή, από την οποία θα μπορούμε να αντιλήσουμε διδάγματα. Επίσης να τονίσω ότι ο ΕΛΚ υπενθύμησε μέσα από τις διάφορες τροπολογίες ότι ζητούμε τον αποκλεισμό των δημοσίων υπηρεσιών από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Ε, τέλος, ε, θα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει τις συζητήσεις για την ισότητα των φύλων στη διεθνή σκηνή, όπως στους κόλπους του ΟΗΕ και του ε, ΠΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στη Συμπρόεδρο, η οποία θα λάβει το λόγο ως ε, συνεισηγήτρια. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν, κυρίως τις δύο συνεισηγήτριες. Εγώ εκφράζω την άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Διαβάζοντας το κείμενο συνειδητοποίησα ότι έχει μια ιδεολογική απόχρωση ε, πολύ συγκεκριμένη. Ε, δεν θέλω η Ευρώπη να γίνει πολύ ακαδημαϊκή και να βγάζει λογίδρια. Δεν λέω ότι γίνεται έτσι τιμωρητική, αλλά τουλάχιστον στυλιτεύει έτσι με το δάχτυλο διάφορες χώρες, οι οποίες δεν έχουν υψηλά πρότυπα σεβασμού των ανθρωπίνων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι, ότι οι εμπορικές ε, επαφές και οι σχέσεις ε, μεταξύ των χωρών δίνουν ευκαιρίες στις γυναίκες που είναι επιχειρηματίες. Γιατί πιστεύουμε ότι το εμπόριο μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει τις γυναίκες. Αυτό σε μια πρώτη φάση. Και φυσικά ε, από εκεί και πέρα μπορεί να τους δώσει και δυνατότητε να κάνουν καριέρα. Με τις τροπολογίες που θα κάνουμε, πιστεύω ότι θα βελτιώσουμε το κείμενο. Εγώ πάντα στη διάθεση σα είμαι. Όσοι με ξέρουν, ξέρετε ότι έχω αυτή τη διάθεση πάντα να συνεργαστώ με αυτό το πνεύμα πνεύμα. Με τις τροπολογίες θα τονίσουμε τις θετικές πτυχές αυτής της διαδικασίας εμπορικής ολοκλήρωσης. Οι επιχειρηματίες γυναίκες είναι όλο και περισσότερες στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και πιστεύω ότι εκείνες εποφελούνται από, τις από τα εμπορικά ανοίγματα. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, κυρίως ειδικά ε, των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που τις διευθύνουν γυναίκες. Υπάρχουν στατιστικές μελέτες που μας ε, εξηγούν ποια είναι η διάσταση του φύλου με πολύ πιο λεπτομερή στοιχεία. Πρέπει να τις λάβουμε υπόψη. Είναι σημαντικό να μελετήσουμε τα στοιχεία, να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα, ούτως ώστε να ξεπεράσουμε τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες. Εγώ είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα συνεργαστούν πολύ καλά οι συγγήτριες, αλλά και οι σκιώδεις συγγητές. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο από τους σοσιαλιστές, η κυρία Νόισλερ. Δεν είναι εδώ. Α, τότε κυρία Ροντρίκες Πινέρο. Ευχαριστώ και τις δύο για τους συμπρόεδρους. Καταρχάς, ζητώ συγγνώμη από την Μαρία Νοέλ, που είναι η σκιώδη εισηγήτρια, δεν μπόρεσε να παραστεί. Μου ζήτησε να, της, να σας πω ποιο είναι το, ποια είναι η άποψή της. Καθώς σας εύχεται καλή επιτυχία. Ευχαριστώ ακόμα τις δύο συνεισηγήτριες, την κυρία Γιώργκ από την Επιτροπή Γυναικών, με την οποία είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πολλές φορές και την Ελεονόρα Φορέντσα. Αυτό το κείμενο έχει συγκεκριμένες ε, προτάσεις για την ε, ισότητα στο εμπόριο και μιλάει για την ανάγκη να βάλουμε ε, δεσμευτικές ρήτρε για τα εργασιακά δικαιώματα, ειδικά σε τομείς όπου δουλεύουν πολλές ε, γυναίκες να λειτουργούν με μεγάλη ευθύνη. Εμείς οι σοσιαλιστές μας ενδιαφέρουν αυτοί οι στόχοι και βεβαίως θα υποστηρίξουμε την κατεύθυνση αυτή. Το υπόλοιπο κείμενο και οι τροπολογίες της ΓΚΟΕ νομίζω επικεντρώνεται υπερβολικά σε μία σειρά από τομείς και κεφάλαια που επηρεάζουν ειδικά αρνητικά τις γυναίκες. Ε, παραδείγματος χάρη γεωργία, ε, δημόσιες προμήθειες, ε, διανοητική ιδιοκτησία. Εγώ διαφωνώ με αυτό και προσωπικά και ως ομάδα. Γιατί για να βάλουμε την διάσταση του φύλου στην εμπορική πολιτική το θέμα δεν είναι να αποκλείσουμε διάφορους τομείς από τη διαπραγμάτευση. Αντίθετα, θα πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα και να πολεμήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση, ούτως ώστε οι γυναίκες να μπορούν να υποφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες. Με τις ίδιες συνθήκες που υποφελούνται και οι άντρες. Και θα ήθελα να πω στις δύο συνεισηγήτριες να το σκεφτούν το θέμα για να φτάσουμε σε μια συμφωνία επ' αυτού. Φυσικά και συμφωνούμε ότι μέχρι στιγμής, όπως λέει και η έκθεση, η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Κομισιόν δεν παρουσίασε σχεδόν καθόλου, δεν έδωσε μάλλον καμία σημασία στο θέμα του φύλου. Όμως λίγο-λίγο άλλαξε αυτή η στάση προς τη σωστή κατεύθυνση, χαίρομαι γι' αυτό και υπό αυτή την έννοια ευχαριστώ όλους όσους ε, έκαναν προσπάθεια για να γίνει αυτή η αλλαγή. Όπως λέει και η έκθεση, είναι αλήθεια ότι η νέα στρατηγική ένα εμπόριο για όλους δεν έχει καμία αναφορά στην ε, γυναίκα και η διάσταση του φύλου στην εμπορική πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην ε, χειραφέτηση των γυναικών. Και σε αυτή πρέπει να βασίζεται, αλλά όχι μόνο. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας το ρόλο των γυναικών ως εργαζόμενες και ως ε, καταναλώτριες, όπως λέει και η έκθεση. Πέρασαν 20 χρόνια από τη δήλωση του Πεκίνου και ακόμα οι γυναίκες είμαστε πάνω από το 70% των ε, δισεκατομμύρια ενδεών ανθρώπων του κόσμου. Δηλαδή, η φτώχεια έχει πρόσωπο και έχει γυναικείο πρόσωπο. Όμως η Κομισιόν διορθώνει τα πράγματα λίγο-λίγο. Στην ε, έκθεση ε, για την εφαρμογή της στρατηγικής για πρώτη φορά αναφέρεται η δέσμευση ότι σε επόμενες διαπραγματεύσεις με αρχές γενομένες από τη Χιλή θα υπάρχει η διάσταση του φύλου και ένα ειδικό κεφάλαιο. Και η, Επιτροπή, η Επίτροπος Μάλστρομ εδώ στην Επιτροπή μας είπε ότι θα υπάρχει ένα κεφάλαιο για το φύλο και την ισότητα του φύλου, των φύλων. Η, το ψήφισμα για την Χιλή ε, ψηφίστηκε με μεγάλη ε, πλειοψηφία. Γι' αυτό λοιπόν μετά από την συντριπτική πλειοψηφία που υποστήριξε αυτή την έκθεση, αυτό το ψήφισμα για τη Χιλή, μου κάνει εντύπωση που το ΕΛΚ δεν θέλει ειδικό κεφάλαιο για, την, για το φύλλο. Σκεφτείτε πώς σκέφτεστε και πώς βλέπετε το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ίσως πρέπει να θεωρήσετε. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι μου φαίνεται σημαντικό να βάλουμε τη δέσμευση, με δεσμευτικό τρόπο, ε, τη διάσταση του φύλου ε, στα θέματα που ρυθμίζει ο ΠΟΕ. Ε, και να μπει ήδη ε, από την ε, διάσκεψη του Buenos Aires το Δεκέμβριο. Και θα πρέπει να είναι εγκάρσια και πολυμερής αυτή η διάσταση. Έχουν γίνει βήματα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι σαφώς ανεπαρκή. Και τώρα θα ήθελα να μιλήσω για τις τροπολογίες που παρουσιάσαμε, που έχουν σαν στόχο να δώσουμε διάφορες αποχρω... διαφορετική απόχρωση και να ενισχύσουμε την έκθεση με θετικές προτάσεις επικοδομητικές. Πώς να δώσουμε νέες ευκαιρίες φερειπίνες στις γυναίκες μέσω της ε, ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής. Από τις 334 τροπολογίες εμείς παρουσιάσαμε τις 106 για να επιτύχουμε δηλαδή αυτόν τον στόχο ακριβώς. Και ελπίζω ότι όλοι οι συγκητές και από τις δύο εμπλεκόμενες επιτροπές θα συμφωνήσουμε όχι μόνο προς το στόχο αλλά και ως προς τα μέσα για να τον υλοποιήσουμε που είναι το πιο σημαντικό. Υπ' αυτή την έννοια δεν νομίζω να, ότι πρέπει να δείξουμε ακαμψία και αδιαλαξία. Αντίθετα κάνω έκκληση να είμαστε συμβιβαστικοί συνενετική. Και να μην ξεχνάμε το στόχο που εδώ και χρόνια δεν μπορούμε να πετύχουμε. Με ένα κεφάλαιο ε, για το φύλλο, το εμπόριο θα είναι πιο αποτελεσματικό. Θα πρέπει να βάλουμε όμως δεσμευτικούς στόχους γι' αυτό. Και αυτό ε, υπάρχει, υπάρχει η τροπολογία 160. Επίσης, στην 275 λένε ότι θα πρέπει να βάλουμε εμπειρογνώμονες άντρες και γυναίκες για θέματα φύλου σε όλες τις φάσεις των διαπραγματεύσεων, ε, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των συμφωνιών. Αυτά τα λέει 275. Επίσης, ζητάμε να υπάρχει μια μεθοδολογία που θα ε, συμπεριλαμβάνει μελέτες με βάση στοιχεία ε, άνα φύλο, άνα τομέα και με δείκτες. θα πρέπει να γίνονται τέτοιε μελέτες και εξ ε, για να δούμε επίσης και πώς θα εφαρμόσουμε μέτρα και μέτρα διορθωτικά της κατάστασης επίσης. Ζητάμε ενεργητικά μέτρα σε μέτρα σε τομεί που έχουν μεγάλη οικονομική επίπτωση στι γυναίκε. Όπω παραδείγματο σε μικρομεσαίε επιχειρήσει, στον ηλεκτρονικό τομέα, στα κλωστοφαντουργικά, στα γεωργικά, διανοητική ιδιοκτησία, γεωγραφικέ ενδείξει για τα γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα. Γιατί και οι γυναίκες της υπαίθρου επηρεάζονται, όπως και οι γυναίκες των πόλεων. Και θα, εντάξει, τελειώνω σύντομα. Είναι σημαντικό να δράξουμε την ευκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που συλλογικά η ΙΝΤΑ και η Επιτροπή Γυναικών θα κάνουμε σε μία ε, έκθεση πρωτοβουλίας το θέμα θα μιλήσουμε για την εμπορική πολιτική και τη διάσταση του φύλου. Το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού περιμένει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι θα πρέπει να αρθούμε στο ύψο των περιστάσεων και των ευθυνών μα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο. Δυστυχώ στι 6.30 ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε την αίθουσα. Ξέρω τον Έρνεστ που είναι καταπληκτικό, τον εκτιμώ, είναι από του πράσινου. Έρνεστ, κατάπληξε με. Σε πολύ λίγα, σε δύο λεπτά. Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ε, δύο ε, για ένα πολύ καλό κείμενο, ε, το οποίο νομίζω πως ε, καλύπτει αυτό το πρόβλημα του ότι δηλαδή η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τελευταία χρόνια υπήρξε τελείως τυφλή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα φύλου. Και ήρθε ο καιρός να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα θα ήθελα να συντομία να αναφερθώ στις τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Σε ό,τι αφορά αυτή την απουσία ε, τη της διάστασης του φύλου από τις αξιολογήσεις αντικτύπου Μα απασχολεί αυτό το ζήτημα και το αναφέρουμε στι τροπολογίε μα και επίση αναφέρουμε ότι για την υπογραφή μια τέτοια ε, συμφωνία ε, χρειαζόμαστε μια κατάλληλη αξιολόγηση αντικτύπου σε ό,τι αφορά το φύλλο και επίση θα πρέπει εμπειρογνώμονε πάντοτε να συμμετέχουν σε αυτήν τη σχετική αξιολόγηση. Και επίση θα πρέπει να υπάρχουν κεφάλαια σε ό,τι αφορά την ισότητα μεταχείριση των φύλων. νομίζω πω αναφέρθηκε σε αυτό η Επιτροπή, δηλαδή περίπτωση ενό τέτοιου κεφαλαίου στο πλαίσιο τη διαπραγμάτευση συμφωνία με τη Χιλή και νομίζω πω αντίστοιχο θα πρέπει να συμβαίνει σε σχέση με όλε τι συμφωνίε, δηλαδή πάντοτε. Επίση, θα θέλαμε να υπάρχει και ένα focal point σε ό,τι αφορά το φύλλο, πάντοτε δηλαδή στα πλαίσια τη Ελληνική Διευθύνση Εμπορίου και επίση θα θέλαμε να έχουμε αποκεντρωμένα ε, ε, δεδομένα ε, και συγγνώμη, αθρηστικά σωρευτικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φύλλου, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μια αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τι υφιστάμενε συμφωνίε και το πώ αυτέ έχουν επιπτώσει στι γυναίκε. Υπάρχουν και μια σειρά από περαιτέρω προτάσει που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά θα ήθελα να να είμαι σύντομο εδώ στην παρέμβασή μου. Έχουμε και άλλε ιδέε και είμαστε ε, βέβαια διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τι δύο συνεισηγήτριε, ούτω ώστε να φάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν, αν ξέρετε του συναδέλφου, ξέρετε πόσο καλέ είναι. Τώρα, ε, Λίδια Άντερσον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα δίνω το λόγο για ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη. Όχι πάνω από ένα λεπτό. Uh, like Σας ευχαριστώ. Ε, Ζήτω συγγνώμη εκ μέρου τη επακεφαλή τη ε, μονάδα μα, ε, τη η οποία βρίσκεται αυτή την περίοδο και συζητά το κεφάλαιο σε ό,τι αφορά το όλο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή σας ε, και την Επιτροπή ΦΕΜΕ σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη αυτής της διάσταση του φίλου στην μια ε, πολιτική και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες εργασίες ε, που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εφαρμογή της στρατηγικής του εμπορίου για όλους αλλά και τη στρατηγική της Ένωσης σε ό,τι αφορά το Aid for Trade, δηλαδή βοήθεια για εμπόριο, αλλά και την πρόσφατη μελέτη που άρχισε να εκπονεί η Επιτροπή. Όλα αυτά δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν στη διάσταση του φίλου. Επίση, το ζήτημα ζήτημα των δικαιωμάτων ε, τη γυναίκα έχουν αρχίσει να περιλαμβάνονται στι διαπραγματεύσει, αλλά ε, τα ε, δεδομένα διαφοροποιημένα αναφύλλω ε, δεν υπάρχουν ακόμα. Αυτό δηλαδή παραμένει μια πρόκληση. Επίση, στα σχετικά κεφόλαια εμπορίου και βιώσιμη ανάπτυξη αναφερόμαστε στι συμβιβάσει του ILO, δηλαδή του Διεθνού Οργανισμού Εργασία, ό,τι αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ των δύο φύλων. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτέ οι διατάξει, ειδικότερα σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου με οικογένειε, δεν έχουν ακόμα υπογραφεί από όλε τι συμμετέχουσε χώρε. Επίσης, Κλείνοντα να πω ότι όπω αναφέρθηκε, υπάρχει ανάγκη για περισσότερα δεδομένα για περισσότερη έρευνα σε σχέση με αυτή τη διάσταση και έχουμε προβλέψει μια ε, ε, νέα μελέτη σε ό,τι αφορά τον τρόπο συλλογή ε, περαιτέρω δεδομένων σε ό,τι αφορά τον όρο των γυναικών και την απασχόληση των γυναικών, όπω δηλαδή είχε προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, έχουμε ξεκινήσει εργασίε από αυτού του ζητήματο με άλλου διεθνού οργανισμού και θα εργαστούμε ε, στο πλαίσιο δηλαδή της εξοργανωμένης συμφωνίας ε, με τη Χιλή επί αυτού του κεφαλαίου ε, για, το φύλλο και ε, βέβαια αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε το ποια συγκεκριμένα ζητήματα θα καλυφθούν. Και τέλος, ναι, θα ήθελα να πω ότι αξιοποιούμε κάθε δυνατή ευκαιρία ούτω ώστε να προβούμε σε περισσότερη ευαισθητοποίηση για αυτά τα ζητήματα. Για παράδειγμα, διεθνώ μέσω τη υποστήριξη μια δήλωση σε ό,τι αφορά το empowerment, δηλαδή την απόδοση, αν θέλετε, αυτεξουσιότητα τη γυναίκα και σε οικονομικό και σε επίπεδο απασχόληση και στο πλαίσιο τη διάσκεψη κορυφή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου αυτό το Δεκέμβριο στον Πουένο Άρη. Σα ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και τώρα μια πολύ σύντομη καταληκτική παρέμβαση από την συγκεκριμένη κυρία Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεισφορά της, τη τελευταία της παρέμβαση. Ευχαριστώ εκ νέου τους και όλους που πήραν το λόγο, είτε στα πλαίσια της Επιτροπής ΙΝΤΑ, είτε στα πλαίσια της Επιτροπής ε, ΦΑΜ. Θα ήθελα τηλεγραφικά να σας πω ότι το γεγονός ότι χαρακτηρίζουμε ε, ιδεολογική αυτή την έρη είναι μια κλασική προσέγγιση. Η βάση αυτής της έκθεσης είναι ότι το εμπόριο πρέπει να συνεισφέρει όχι στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά στην κατάργηση των ανισοτήτων αυτών. Τι είναι αυτό, είναι ιδεολόγημα. Νομίζω ότι είναι μια αρχή που μου βρίσκει όλους σύμφωνους, ό,τι απόψεις και να έχουμε. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά. Thanks uh, to my co-chair. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και στη συμπρόεδρό μου. Νομίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε στις 24 Ιανουαρίου και θα εξετάσουμε την ε, έκθεση. Ευχαριστώ.